Hello everyone. If there are no Αν δεν έχετε αντίρρηση, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη χωρίς τροποποιήσεις. Προβλέπεται μία δημόσια ακρόαση με συμμετοχή της ΕΜΒΗ σε σχέση με τους ενδοκρινικούς ε, καταράκτες στις 22 Μαρτίου από τις 10 ε, παρατέταρτο και όλοι καλείστε να συμμετάσχετε. Στις 27 Μαρτίου από τις 2 το μεσημέρι θα γίνει ένα εργαστήριο της Επιτροπής για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα για τα βαρέα οχήματα και τα μικρά φορτηγά. Ε, καλείστε όλοι και ε, στις 12 Απριλίου θα, δεν θα γίνει η απογευματινή συνεδρίαση, έχουν γίνει ορισμένες αλλαγές. Ο κύριος Ματώ Μενεγκάτη που προέρχεται από τη νομική υπηρεσία θα ε, βρίσκεται πλέον μαζί μας. Σας καλωσορίζουμε για σήμερα. Έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσες και όπως ξέρετε Η συνεδρίασή μας μεταδίδεται απευθείας στο διαδίκτυο. Το πρώτο θέμα είναι οι κοινοί κανόνες για ορισμένες συνδεδευμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών. Ο κύριος Νταντά είναι ο εισηγητής, ο οποίος έχει και το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σήμερα στην Ευρώπη οι οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 49% του συνόλου των μεταφορών εμπορευμάτων και ο πολυτροπικός, οι πολυτροπικές μεταφορές είναι το 12%. Οι μεταφορές μέσω σιδηροδρόμου είναι περίπου 19%, ενώ οι μεταφορές με ναυσιπλοεία είναι το 6,4%. Χρήσιμο είναι λοιπόν να υπενθυμίσουμε δύο ορισμούς. Ποια είναι η συνδυασμένη μεταφορά και ποια είναι η πολυτροπική μεταφορά. Η πολυτροπική μεταφορά είναι η διαμετακόμιση εμπορευμάτων η διαδοχική, ενώ η συνδυασμένη μεταφορά είναι μία από, ε, ένας από τους πολυτροπικούς ε, τρόπους μεταφορών και διέπεται από την οδηγία 92-106 που θέλει η Επιτροπή να αναθεωρήσει σήμερα. Γιατί η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενδιαφέρεται για αυτά τα κείμενα. Γιατί ε, το εμπόριο, μεταφο... Ε, το... οι μεταφορές των αγαθών θα αυξηθούν πάρα πολύ μέχρι το 2050 με την οικονομική ανάπτυξη, με την επιστροφή στην ανάπτυξη. Έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση από βαρέα οχήματα. Η συνδυασμένη μεταφορά λοιπόν παρουσιάζει πολλά πλέον εκτήματα. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 81% των πολυτροπικών μεταφορών είναι διασυνοριακές και έτσι οι υποδομές αυτές μπορούν να βοηθήσουν ε, ζώνες που ε, είναι ε, σε μειονεκτική θέση, όπως είναι οι πολλές, πολύ ορεινές περιοχές ή να αποσοβηθεί και να μειωθεί ο σεισμογενής κίνδυνος, γιατί όταν θα φύγουν τα πολλά οχήματα μεταφοράς αγαθών από τους δρόμους, η πίεση προς τα εδάφη θα είναι μικρότερη. Οι 25 χρόνια έχουν περάσει από τότε που τέθηκε σε ισχύ η προηγούμενη οδηγία. Σήμερα τα διακυβεύματα είναι πολλά. Έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες στην Ευρώπη να αυξήσουμε την πολυτροπική μεταφορά και πρέπει ε, να αυξήσουμε τις επενδύσεις στους εμπορευματικούς σταθμούς διαμετακόμισης των εμπορευμάτων. Είναι άνηση και η εφαρμογή, άνηση και ελληματική η εφαρμογή της οδηγίας από τα κράτη-μέλη, δεν είναι πολύ σαφής η οδηγία και έτσι το κάθε κράτος μέλος την ερμηνεύει διαφορετικά. Υπάρχουν διαρθρωτικές ανισότητες και ε, δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να είναι ανταγωνιστικά, ορισμένα από αυτά. Σε κάθε περίπτωση οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, καλύπτουν κάποια από τα σημερινά κενά και ελλείμματα. Έχω τρεις βασικές ομάδες τροπολογιών να προτείνω. Πρώτον, μέτρα στοχευμένης στήριξης. Δεύτερον, βελτίωση της αλυσίδας των logistics χάρη στη νέα τεχνολογία. Και τρίτον, εναλλακτικά καύσιμα στις συνδυασμένες μεταφορές ως προς τα στοχευμένα μέσα στήριξης. Στόχος της Κομισιόν είναι ανά 300 χιλιόμετρα παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση να Έχουμε αυτή τη γεωγραφική λογική της ε, εναλλαγής. Κάθε 300 χιλιόμετρα να αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρονται τα εμπορεύματα για να μειώνεται το βάρος στο περιβάλλον. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να διατηρήσουμε μόνο το γεωγραφικό κριτήριο, αλλά και άλλα κριτήρια. Και θα πρέπει τα μέσα στήριξης να είναι στοχευμένα καλύτερα. Να έχουμε επενδύσεις στους σταθμούς ε, διαμετακόμισης εμπορευμάτων, στον εξοπλισμό, στις νέες τεχνολογίες, αλλά και επενδύσεις στην κατάρτιση του εργασιακού δυναμικού. Να ενθαρρύνονται οι επενδύσεις και οι χρηματοδοτήσεις στις διασυνοριακές δραστηριότητες, ειδικά στις ορεινές περιοχές, όπου η μεταφορά είναι πολύ πιο δύσκολη. Τώρα, Δεύτερη ομάδα τροπολογιών για τις νέες τεχνολογίες. Να ενθαρρύνουμε την προσφυγή σε αυτές τις νέες τεχνολογίες, τη συστηματική ψηφιοποίηση των δεδομένων για να είναι πιο αποτελεσματικές οι δράσεις οι μεταφορικές και να μειωθεί το κόστος τους. Τρίτον, τις τροπολογίες για το εναλλακτικό καύσιμο. Ούτως ή άλλως η οδηγία θέλει να μειώσει την επίπτωση που έχει η μεταφορά των εμπορευμάτων στον περιβάλλον. Και αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος της συνθήκης των Παρισίων και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για το κλίμα για το 2030. Η οδηγία δεν προβλέπει μέσα στήριξη για τα οχήματα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα. Όμως το ε, τα εμπορεύματα κατά 5% μεταφέρονται με φορτηγά και τα φορτηγά κατά 95% εξαρτώνται από το αορυκτά καύσιμα. Εμείς προτείνουμε εναλλακτικά καύσιμα, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός, τρόπος καύση στο κινητήρα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα και θέλουμε να στηριχθούν αυτά τα μέσα. Από εκεί και πέρα. Για το καμποτάζ, γιατί υπάρχουν πολλοί τέτοιοι φόβοι, δίδεται παρέκκληση από τον κανόνα του καμποτάζ στις συνδυασμένες μεταφορές. Βεβαίως αυτός ο κανόνας δεν ισχύει για τις εθνικές μεταφορές και δεν θα πρέπει να οδηγήσει τελικά στην de facto κατάργηση του καμποτάζ. Σε κάθε περίπτωση οι εμπορευόμενοι, οι οικονομικοί συμμετέχοντες στην αγορά είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό πρέπει το, η γραφειοκρατία να είναι όσο το λιγότερη. Είμαι στη διάθεσή σας, θα ακούσω όλες τις τροπολογίες που... και θα τις δεχτώ με μεγάλη ευχαρίστηση και θα συναντήσω το συντομότερο δυνατό τους όδης εισηγητές για να προετοιμάσουμε τη συνέχεια που θα δοθεί στο έργο μας. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή τον κύριο Τανασέσκου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ξέρετε, προσπαθούμε να μειώσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο των ε, μεταφορών και αυτό είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους. Το Μάιο 2017 το η Europe on the Move μίλησε για μία μετάβαση σε καθαρή κινητικότητα με ένα πρώτο πακέτο προτάσεων. Η αναθεώρηση του κανονισμού 92 κάθετος 106 κάθετος ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ε, μέρος αυτού του δεύτερου πακέτου μεταφορών. Και οι συνδυασμένες μεταφορές είναι το μόνο νομικό μέσο έτσι ώστε να περάσουμε από τις οδικές μεταφορές σε μεταφορές με χαμηλότερη με χαμηλότερες εκπομπές και επίσης να περάσουμε από τις οδικές σε άλλα μέσα, άλλες μορφές μεταφορών. Οι συνδυασμένες μεταφορές είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντισταθμίσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο των μεταφορών, αλλά θα πρέπει να εξελίξουμε και ολόκληρο το δυναμικό μας. Η πρόταση της Επιτροπής μας δίνει διασαφηνίσεις για την εφαρμογή σε επίπεδο κρατών μελών. Επίσης, η πρόταση της Επιτροπής μιλά για την επέκταση οικονομικής υποστήριξης για όλες τις συνδυασμένες μεταφορές μέσα στα πλαίσια και των διατροπικών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί μίλησε για νέα γεωγραφικά κριτήρια τα οποία όμως δεν έχουν καμία σχέση με τα τερματικά, γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα των ε, εμπορικών ροών. Η οδηγία 92 κάθετος 106 κάθετος ε θα πρέπει να λάβει υπόψη την ειδική νομοθεσία στον τομέα των μεταφορών ενέργειας, περιβάλλοντος και υγείας περιμένω υποδείξεις σας και ελπίζω να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Τόβατς. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάντα γιατί τόνισε για το, τη δυναμική πορεία συνδυασμού μέσων ε, μεταφοράς και μιλάμε και για τους στόχους των Παρισίων ως προς την Συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να μειώσουμε το ε, ανθρακικό, το αποτύπωμα του άνθρακα στον τομέα των μεταφορών και θα δούμε πώς θα μπορέσουν να εξελιχθούν και οι επενδύσεις σε αυτό το τομέα άκουσα και άλλες και διάβασα και άλλες εκθέσεις της Επιτροπής και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν. Αν δείτε το σύστημα συνδυασμένων μεταφόρων σε ευρύτερο πλαίσιο, τότε βλέπετε ότι οι συνδυασμένες μεταφορές σε ένα καλό περιβαλλοντικό πλαίσιο εξαρτάται από, από τους δύο ε, ποταμούς, δηλαδή τον Ρήνο και τον ε, Δούναβη και κατά πόσο απορροφούν δηλαδή τους ε, ρήπους. Και εάν δεν υπάρχει σωστή συμμόρφωση, το Οπότε η διάρθρωση του δικτύου, ιδιαίτερα του σιδηροδρομικού, δεν είναι καθόλου ε, καλή. Και γι' αυτό περνάμε στις οδικές μεταφορές όταν δεν είναι καλό το σιδηροδρομικό δίκτυο. Όταν δείτε ε, λοιπόν τη μετάβαση στις οδικές μεταφορές θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μία εξέλιξη των τελευταίων 20-30 ετών. Ε, όταν πάω πίσω στα παιδικά μου χρόνια, βλέπω ότι οποιαδήποτε ε, εταιρεία είχε αποθηκευτικούς χώρους και οι μεταφορές σε αυτούς τους αποθηκευτικούς ε, χώρους δεν είχε σημασία ως προς το χρονισμό της γιατί υπήρχε μεγάλη χωρητικότητα. Από την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 90 και μετά το 2007 βλέπετε σαφώς ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ε, απαλλαγούν από τους αποθηκευτικούς χώρους ή τους μειώνουν. Και φτάσαν σε ένα εφοδιαστικό σύστημα όπου ο χρονισμός ε, παίζει μεγάλο ρόλο. Αν θέλω ένα εξάρτημα για το αυτοκίνητο τότε θα πάω στο συνεργείο της γειτονιάς και θα στείλει ένα mail σε ένα κέντρο ε, εφοδιαστικής, εκατοντάδες χιλιόμετρα ίσως μακριά και ίσως το εξάρτημα να έρθει αεροπορικός ή με κάποιο άλλο τρόπο. Και επειδή ο παράγων χρονισμός είναι πολύ σημαντικός, τότε θα, μάλλον θα φτάσει μέχρι εμένα ο δικός. Άρα, αν δεν λάβουμε υπόψη τους αποδικευτικούς χώρους, δεν θα κάνουμε, δεν θα φτάσουμε και με, σε μεγάλες διαφορές. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι κρίσιμο και χάρηκα πολύ που συνεργάστηκα με τον εισηγητή. Ευχαριστούμε κύριε Τροβάλτσα. Οι ή οι άλλε σκιώδεις εισηγητές δεν είναι εδώ παρόντες. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Αν όχι, λοιπόν, από την Επιτροπή Έχουμε τον κύριο Σανταμάτο μαζί μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για το σχέδιο εκνομοδότηση αυτό και να πω ευθύ εξ αρχή ότι η μεγάλη πλειονότητα των τροπολογιών κινούνται στην κατεύθυνση των όσων και εμείς προσπαθούμε να πετύχουμε με την πρόταση αυτή. Άρα θεωρούμε ότι είναι ευπρόσδεκτες από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διευκρινίζουν αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Τρία βασικά ζητήματα είναι τα, τα ζητήματα τα οποία αναφέρονται σε ό,τι αφορά το καμποτάζ και το σχετικό waiver. Η ερμηνεία είναι ίδια με αυτήν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι αυτή η απαλλαγή θα πρέπει να ισχύει μόνο για τις συνδυασμένες διασυνοριακές μεταφορές. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της ενθάρρυνσης και της παρότρινσης και προώθησης καθαρών οχημάτων, είναι μια ιδέα την οποία εν γέννη υποστηρίζουμε. Ενδεχομένω να υπάρχουν δυσκολίε που θα αντιμετωπίσουμε, να δούμε πώ θα ενταχθεί αυτό στο πλαίσιο της πρότασης Ίσως ε, ο σκοπό είναι λίγο διαφορετικό ε, Ελαχιστοποίηση των οδικών μεταφορών για να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα τη ε, της κυκλοφοριακής Αλλά ενδεχομένω να μπορέσουμε να βρούμε και κάποιε ιδέε για την υποστήριξη των καθαρών οχημάτων. Ένα τρίτο ζήτημα το οποίο τονίστηκε σε ό,τι αφορά τα 300 χιλιόμετρα και την ύπαρξη σταθμού κάθε 300 χιλιόμετρα και εμεί συμφωνούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια κάποια ευελιξία. Αυτό αποτελεί μια γενικότερη ενδεκτική, αν θέλετε, στοχοθεσία. Εξαρτάται φυσικά και από τις συγκεκριμένες συνθήκες. Συμφωνούμε ότι δεν μπορεί να ακολουθείτε αυτός ο στόχος ανελαστικά. Κάποια σχόλια τώρα, αν μου επιτρέπετε, για κάποιες συγκεκριμένες ε, τροπολογίες. Οι οποίες ενδεχομένω να παρουσιάσουν πρόβλημα. Για τον πιο κοντινό κατάλληλο σταθμό. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια που θα ορίσουν το σταθμό αυτό στην πρόταση, στο άρθρο 1, παράγραφος 3, σημείο 3, Ήδη έχουμε συμπεριλάβει κάποια τέτοια κριτήρια και θεωρώ ότι χρήσιμο θα ήταν να παραμείνουν στο διεκτακτικό αυτά τα, κριτήρια και όχι σε πράξεις κατά εξουσιοδότηση, επιτελεστικές πράξεις για το θέμα του να καταστεί υποχρεωτικό για τα κράτη-μέλη να αποδεχτούν τη χρήση του του σταθμού. Αυτό όντως το επιθυμεί διακαώς ο κλάδος αλλά θεωρώ ότι πολύ πολύ δύσκολο θα περάσει από το Συμβουλίο. Κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. Εδώ η συμμόρφωση με τους σχετικούς εθνικούς κανόνες θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε περίπτωση. Και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμπεριληφθεί στην πρόταση μια απαλλαγή για την υποχρέωση κοινοποίησης. Γιατί οι κανόνες αυτοί ισχύουν οριζόντια για διάφορους ε, τομείς. Δεν θεωρούμε ότι θα είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί μία συγκεκριμένη διάταξη Τέλος, γίνεται μία αναφορά στην τροπολογία 3 για τις ε, συνθήκες εργασίας και τις κοινωνικές συνθήκες. Φυσικά, είναι σε φάση ε, οι συνθήκες για τον κλάδο, αλλά η εναρμόνιση μεταξύ των διάφορων τρόπων μεταφοράς δεν είναι κάτι το οποίο στην παρούσα φάση είναι άμεσο. Και σε ό,τι αφορά την τροπολογία 19, να κοιτάξουμε λίγο τη διατύπωση, αν θέλετε, γιατί συμφωνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, επιτελεί τα καθήκοντά της ως θεματοφύλακα των συνθήκων, αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ε, αρμόδια και υπεύθυνη για την καταλληλοποίηση της οδηγίας. Αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και εδώ λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μικρή προσαρμογή. Στο σημείο αυτό θα κλείσω και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ λέει και Πρόεδρος. Ο κ. Νταντά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις των συναδέλφων που πήραν το λόγο. Πιστεύω ότι θα κάνουμε πολύ καλή δουλειά μαζί. Άκουσα και με πολύ προσοχή τις αντιρρήσεις και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να το συζητήσουμε. Είμαστε εδώ για να προτείνουμε, για να νομοθετήσουμε και όχι για να ακολουθούμε πάντοτε κατά γράμμα τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ολοκληρώνεται η εξέταση αυτού του σημείου της ημερήσιας διάταξης. Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών 11 Απριλίου στις 11 το πρωί. Και ψηφίζουμε στην Επιτροπή μας στις 16 ή στις 17 Μαΐου. Προχωρούμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επεξεργασία των λιμάτων στις αστικές περιοχές. Έχουμε την κυρία Μανφρέντι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, τον κύριο Ματίας Μαλγκάη, αν προφέρω σωστά το όνομά σας, επικεφαλής της μονάδας του τμήματος του Αρμοδίου. Θα ξεκινήσουμε δίνοντάς σας το λόγο για 10 λεπτά και μετά τα κράτη-μέλη θα θέσουν τις ερωτήσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς και όλα τα μέλη για το ενδιαφέρον που τρέφουν για αυτή την εργασία και κυρίως ε, για ε, την έκθεση που θα παρουσιάσω εντός ολίγου. Έχω μία μικρή παρουσίαση για να δείξω τον, ε, το επίπεδο συμμόρφωση με την ειδηγία, τον αντίκτυπο στο περιβάλλον, τι κάνουμε για τα θέματα της εφαρμογής αλλά και για τα συμπεράσματα που αντλούμε να εξηγήσω δύο-τρεις όρους για όσους δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι ε, με το θέμα. Έχουμε την έννοια του population equivalent, αντίστοιχο στο πληθυσμό. Ποιοι είναι οι στόχοι στις πόλεις και ε, στους ε, τόπους. Έχουμε αστική περιοχή όταν έχουμε πάνω από 2.000 άτομα υποχρέωση να συλλέγονται τα λίματα όταν έχουμε ε, τοπικές κοινότητες με, με αντίστοιχο πληθυσμό population equivalent άνω του 2.000 ατόμων και υποχρέωση να επεξεργαστούμε τα ε, λίματα. Είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί, δεν θέλουμε καθόλου να χρησιμοποιούμε όρους η Ευρώπη των 15, η Ευρώπη των 30 και ούτω καθεξής επειδή υπήρχαν διαφορετικές προθεσμίες λόγω της διαφορετικής ημερομηνία κατά την οποία προσχώρησαν οι διάφορες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, γι' αυτό ε, ομαδοποιούμε τις χώρες με αυτόν τον τρόπο. Πρόσφατα, ε, η Επιτροπή δημοσίευσε την ένατη έκθεση εφαρμογής μετά από 16 χρόνια από τότε που δημοσιεύθηκε η πρώτη έκθεση για να σας δώσω μια βασική ιδέα για το μέγεθος του εγχειρήματο. Έχουμε εξετάσει 23.500 ε, κοινότητες, πόλεις, κομοπόλεις. Η οδηγία ισχύει και εφαρμόζεται για 604 εκατομμύρια σε αντιστοιχεία πληθυσμού, ΠΕ δηλαδή, population equivalent, σε ε, περίπου 500 και μεγάλες πόλεις. Τώρα δύο πολύ βασικές έννοιες που θα δείτε, ορολογίας. Δύο διαφορετικοί είναι οι τρόποι να εξετάσουμε πώς εφαρμόζεται η οδηγία σε κάθε κράτος μέλος. Στο πάνω μέρος της οθόνης, στον πάνω πίνακα, βλέπετε το ποσοστό συμμόρφωσης βάσει της νομικής μεθοδολογίας που χρησιμοποιούμε και την οποία επικύρωσε το δικαστήριο. Δηλαδή, όταν βλέπουμε πότε πότε εφαρμόζεται πλήρως η οδηγία. Άρα άμα αποτυχάνει κάποιος Δήμος να την εφαρμόσει σε ορισμένες πτυχές της παίρνει 0%, αν την εφαρμόζει πλήρως παίρνει 100%. Και άρα εδώ βλέπετε τις χώρες όπου η οδηγία ισχύει για πάρα πολλά χρόνια φτάνουν στο 100% της εφαρμογής σε ό,τι αφορά τη συλλογή των λιμάτων και είναι η πρώτη στήλη και αρκετά ψηλά, περίπου στο 90% ε, εφαρμόζουν τη δευτερογενή επεξεργασία αλλά και την πιο αυστηρή επεξεργασία. Αυτά στην παλιά Ευρώπη των 15 να το πούμε έτσι. Άλλες 13 χώρες έχουν αρκετά ψηλά ποσοστά αλλά όχι ακόμα αρκετά ικανοποιητικά. Αλλά είναι γιατί άρχισε να ισχύει η οδηγία σε αυτές τις χώρες αργότερα, γιατί προσχώρησαν αργότερα. Τώρα, το ποσοστό του νερού που συλλέγεται και υφίσταται επεξεργασία φαίνεται στον κάτω πίνακα και εδώ τα νούμερα απέχουν πολύ από το στόχο. Είναι κάπως καλύτερη εικόνα στους περισσότερους τομείς της εφαρμογής, αλλά είναι ανησυχητικά χαμηλή η εφαρμογή της εκ νέου επεξεργασίας ε, με αυστηρό τρόπο. Μόνο σε 13 χώρες γίνεται αυτό. Τώρα, ένας άλλος τρόπος να εξετάσουμε τη συμμόρφωση με την οδηγία και την εφαρμογή της στα κράτη-μέλη. Να σας δείξουμε τη γεωγραφική κατανομή. Στα αριστερά, με μπλε βλέπετε τις καλές επιδόσεις, τις χώρες όπου ισχύει η οδηγία σχεδόν 100% σε ό,τι αφορά τη συλλογή και δεξιά αυτό που είχαμε πριν, δηλαδή μια εικόνα που μας ανησυχεί πολύ περισσότερη, περισσότερο όταν μιλούμε για τη σωστή επεξεργασία, την πιο αυστηρή και πιο χρήσιμη επεξεργασία. Εδώ σας δείχνουμε κάποιες τάσεις που προσπαθούμε να συλλέξουμε και να διαμορφώσουμε, να απεικονίσουμε δηλαδή. Φαίνεται δηλαδή ότι η κατάσταση βελτιώνεται, η κάτω γαλάζια γραμμή δείχνει μία δυναμική πορεία τώρα με ένα στιγμιότυπο, στατικό απεικόνησης δεν μπορείτε να το καταλάβετε όμως η γαλάζια γραμμή δείχνει ότι 13 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκαναν αυτές τις τεράστιες επενδύσεις για να μπορούν να συλλέ, όχι μόνο να συλλέγουν τα λίματα αλλά και να τα επεξεργάζονται σε βάθος και σωστά. Τώρα, όσοι ενδιαφέρονται σε μεγαλύτερο βάθος, βλέπετε ότι οι τάσεις έχουν μειωθεί. Ε, υπάρχει μια μικρή πτώση εκεί πάνω δεξιά. Η πτώση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι τώρα καταφέρουμε να, να συλλέγουμε καλύτερα δεδομένα και να έχουμε πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ελαφρά τάση μείωσης παροδική. Τώρα, το πιο σημαντικό ο πιο σημαντικός λόγος γιατί το κάνουμε όλο αυτό, γιατί η οδηγία έχει ένα πολύ θετικό αντίκτυπο και στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου. Εδώ σας δείχνουμε κάποιες γραφικές παραστάσεις, δύο τρόπους ερμηνείας του φαινομένου. Ε, βελτιώνεται η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης και Έχουμε παραμέτρους για να ξέρουμε και να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, άρα η εφαρμογή της οδηγίας για την συλλογή, την επεξεργασία, τη διαχείριση των αστικών λιμάτων ε, έχει τεράστιο θετικό αντίκτυπο στην οδηγία ε, για τα ύδατα κολύμβησης και στην ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Και εδώ κάτω έχουμε την βιολογική ζήτηση σε οξυγόνο, είναι μια ένδειξη της οργανικής ρήπανσης της οργανικής μόλυνσης του νερού. Ε, συνήθως όταν υπάρχει αυτή η ζήτηση πολύ, το BOD όπως το λέμε, Biological Oxygen Demand, αυτό δείχνει ότι ασκείται μεγάλη πίεση στα, ε, στα ύδατα και μειώνεται η ποιότητά τους. Ο θετικός αντίκτυπος στο περιβάλλον και στην υγεία δεν είναι το μόνο σημαντικό. Εξίσου σημαντικό είναι ότι ενισχύεται η κυκλική οικονομία με την συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία των αστικών λιμάτων αφαιρούμε τις επιβλαβείς ιδιότητες των θρεπτικών και των βιολογικών ρηπαντών και σύν της άλλης επαναπροσλαμβάνουμε πολλά από αυτά τα θρεπτικά. Ο φόσφορος ας πούμε είναι ένα πεπερασμένο υλικό και είναι σημαντικό να τον έχουμε ενδογενώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε επίσης ότι πολλές ε, χώρες κάνουν εκ νέου χρήση των επεξεργασμένων αστικών λιμάτων και αυτό είναι αντικείμενο ξεχωριστής νομιθωτικής πρότασης που θα προκύψει από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην έκθεσή μας εξετάζουμε και τις ανάγκες για επενδύσεις. Τα κράτη-μέλη αναφέρουν ποιες είδους επενδύσεις, ποιου είδους επενδύσεις χρειάζονται και σε νέες υποδομές, αλλά και στη διατήρηση και την ανανέωση, ανακαίνιση υφιστάμενων ε, υποδομών και είναι ενδιαφέρουσες οι τάσεις που διαγράφονται. 26 δις ευρώ επενδύσεις ετησίως προβλέπονται από τα κράτη-μέλη κάθε χρόνο για τα επόμενα χρόνια και νέες επενδύσεις κυριαρχούν στην Ευρώπη των 13, στην Ευρώπη των 15 η οι επενδύσεις κυρίως προορίζονται για την ανανέωση των υποδομών. Δηλαδή στις χώρες που προσχώρησαν αργά ε, χρειάζονται νέες επενδύσεις γιατί δεν υπάρχει καθόλου υποδομή. Στις χώρες που είναι παλιά μέλη πρέπει να ανανεωθεί η υφιστάμενη υποδομή. Σχεδιάζεται να, αυτή τη στιγμή να είναι ε, συγχρηματοδότηση με το ποσοστό της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανέρχεται στο 26%, όμως πρέπει όλα αυτά να τα δούμε και στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής ε, περίοδου. 10 δις ευρώ προβλέπονται ε, ως προ, από πλευράς νέας χρηματοδότησης τα επόμενα 10 χρόνια και τεχνική βοήθεια Όλο αυτό δείχνει πόσο τεράστιες είναι οι προκλήσεις για τις χώρες και πόσο πρέπει εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστούμε με τις χώρες, να τις βοηθήσουμε για να μπορέσουν να τα φέρουν σε πέρα σε όλα αυτά τα καθήκοντα και να ε, καταφέρουν να εφαρμόσουν την ε, οδηγία αυτή εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στις χώρες με τα μεγαλύτερα προβλήματα, στις χώρες με το, με το χαμηλότερο ποσοστό εφαρμογής, σε συνεργασία με τους συναδέλφους που είναι αρμόδιοι για θέματα συνοχής. Συνεργαζόμαστε με τον ΟΣΑ, με την Παγκόσμια Τράπεζα, πηγαίνουμε επί τόπου, αξιολογούμε τις ανάγκες και ε, θέλουμε να κάνουμε το παν για να διασφαλίσουμε ότι θα έχει η παρέμβασή μας το θετικό αντίκτυπο που ε, τόσο είναι απαραίτητος. Συμπερασματικά για εμάς που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα εδώ και πολύ καιρό. Οι τάσεις είναι θετικές. Υπάρχουν πολλά καλά νέα. Όμως, αν κάποιος ε, ασχοληθεί με το θέμα μόνο σήμερα, είναι λογικό να ρωτά γιατί έχουμε τόσο τεράστια κενά στην εφαρμογή από τη μία χώρα στην άλλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζει τον ενδιαφέρον της στην στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν όλοι να δρέψουν τα ωφέλη, να μπορέσουν να γίνουν οι βέλτιστες επενδύσεις να μπορέσει να υπάρξει περαιτέρω θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα των υδάτων του περιβάλλοντος να προστατευτεί ακόμα περισσότερο η ανθρώπινη υγεία. Όλα αυτά συνδέονται και με τον στόχο ε, βιώσιμης ανάπτυξης ε, υπαριθμών 6. SDG, Sustainable Development Goals. Ε, όλα αυτά αποτελούν αντικείμενο άσκησης αξιολόγησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γίνεται ε, μια δημόσια διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον έκτο ε, αναπτυξιακό στόχο βιώσιμης ανάπτυξης και περιμένουμε τη συνεισφορά σας και σε αυτή τη διαβούλευση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Με χαρά να απαντήσω στα σχόλιά σας και στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ποιος θα ήθελε να λάβει το λόγο για ερωτήσεις. Η κυρία Γιατομάκη είναι η πρώτη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση. Η έκθεση της Επιτροπής δεν αναφέρεται στα φαρμακευτικά υπολείμματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μόλυνση του περιβάλλοντος. Αυτό συζητήθηκε και στα πλαίσια της ε, στρατηγικής σε σχέση με την ε, μικροβιακή αντίσταση με βάση και το REFIT. Θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς ε, προβλέπει η Επιτροπή για το ζήτημα αυτό. Ο κύριος Νταντέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εισήγηση αυτή. Νομίζω ότι έχουμε μία καλή εικόνα για την επεξεργασία του νερού, ιδιαίτερα των λιμάτων νερού, όπως ορίζει η οδηγία. Πώς αντιλαμβάνεται το θέμα η κοινή γνώμη. Τα τελευταία 30 χρόνια αλλάζουμε συνέχεια τα δεδομένα, διότι Στόχος είναι να βελτιώσουμε γιατί οι τεχνολογίες ανάλυσης έχουν βελτιωθεί και έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα πιο ακριβές θερμόμετρο. Η κοινή γνώμη όμως έχει την εντύπωση ότι παρά τις επενδύσεις μας τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα έπρεπε. Θα έπρεπε λοιπόν σε τακτά χρονικά ε, διαστήματα να δημοσιεύουμε και τα τρία βαρόμετρα, διότι αυτά κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση και δείχνουν ότι οι περιβαλλοντικές επενδύσεις, για αυτές τις επενδύσεις χρειάζεται χρόνος για να αποδώσουν. Και ε, γιατί δεν μιλάμε μόνο για μία μονάδα επεξεργασίας λιμάτων, αλλά για ένα γενικότερο πλαίσιο και περιβάλλον που χρειάζεται 5 με 10 χρόνια, έτσι ώστε να αποδώσει και να φανούν τα αποτελέσματα. Νομίζω λοιπόν ότι η κοινή γνώμη δίνει μεγάλη σημασία στο θέμα των υδάτων και θα πρέπει να βελτιώσουμε και την ε, επικοινωνιακή μας πολιτική. Γιατί έχουμε ε, και ένα πρόγραμμα στα σκαριά για τα φαρμακευτικά υπολείμματα και το θέμα των ορμονών, το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και χρειάζεται πολύ χρόνο και χρήμα και γι' αυτό ακριβώς ε, θα πρέπει οι επιστήμονες να ασχοληθούν μακρόν με τις νέες τεχνολογίες επί του θέματος. Ο κύριος Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ. Ακούσαμε την Επιτροπή και δεχόμαστε τα αποτελέσματα που μας προανέφερε, γιατί υπάρχει μία απτή ε, βελτίωση με βάση αυτή την οδηγία. Όμως στην Ιταλία έχουμε μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με το, ε, τον βιολογικό καθαρισμό γιατί υπάρχουν ε, τρεις διαδικασίες επί παραβάση ενώπιον του δικαστηρίου όπου η απόφαση αφορά τους οικισμούς που δεν διαθέτουν βιολογικό καθαρισμό και εκεί όπου δεν υπάρχει επεξεργασία λιμάτων. Άρα οι Ιταλοί πληρώνουν, μάλλον ε, επομίζονται ένα κόστος χωρίς ε, να υπάρχει αντίκρισμα. Στην Ισπρά μαθαίνουμε ότι η ανάκτηση ηλίως δεν χρησιμοποιείται ως ε, λίπασμα γιατί θα είχε μεγάλη θρεπτική αξία για τις γές, αλλά δυστυχώς ε, μεταφέρονται σε χωματερές, κάτι το οποίο δεν οδηγεί σε μία πραγματική επεξεργασία και οικονομίες για τον πολίτη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ανάκτηση της ηλίως που προέρχεται από την δευτερογενή επεξεργασία και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο θα σταθεί περισσότερο στις ευθύνες των τοπικών και περιφερειακών αρχών επί του θέματος. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαρπίρικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ την ίδια ερώτηση έχω να κάνω όπως ο πρώτος Πριν από κάποιο καιρό είχαμε ένα συνέδριο εδώ με το Συμβούλιο Διαχείρισης Υδάτων και από την Ολλανδία και το θέμα των αντιβιωτικών και των υπολοιμμάτων αντιβιωτικών τέθησε σε ό,τι αφορά τα λίμματα από τα νοσοκομεία. Πώς θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν το θέμα αυτό. Κοιτάμε λοιπόν πώ μπορούμε να καταθέσουμε σχετικέ τροπολογίε. Ο τελικό ο τελευταίος ομιλητή, θεωρώ ότι ήταν ε, πολύ ενδιαφέρον γιατί μίλησε και για τέτοιε θρεπτικέ ουσίες κτλ. Αυτό ακριβώ περιλαμβάνει η τελευταία τροπολογία για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Την καταψηφίσατε όλοι όμω, σε ό,τι αφορά και την άποψη του Συμβουλίου Διαχείρισης Υδάτων. Η λύση που είχε προταθεί λοιπόν ήταν αυτή. Να μα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θυμάται πώς έχουν ακριβώς ε, τα πράγματα. Από πολιτικής άποψης όμως ε, έχουν το θέσιο αυτό το πράγμα, ότι σε πολλές περιπτώσεις μιλάμε για το θέμα των υδάτων, αλλά διαπιστώνω ότι στο κοινοβόλιο ψάχνουμε λύσεις ε, σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υδάτων, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς σε κάθε περίσταση ποιος άλλος ασχολείται με τέτοια ζητήματα. Και αυτό ήθελα να το επισημάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ το ίδιο έχω να πω. Τις ίδιες ανησυχίες έχω με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Μισελ Τοντά. Την ερώτηση λοιπόν που ήθελα να θέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τα αστικά αλήματα. Αλλά για να ξαναβρεθούμε σε μια ικανοποιητική κατάσταση σε ό,τι αφορά τα νερά ενός ποταμού, δεν σημαίνει ότι παρόλα αυτά τα έδωτα δεν θα έχουν τοξικές ουσίες. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξή ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως τώρα δεν έχουμε λάβει υπόψη τις ε, μελέτες και τις έρευνες ε, τοξικολογίας. Μπορεί, για παράδειγμα, να έχουμε προβεί σε σωστές δράσεις για να ποταμώσουμε ό,τι αφορά τη βιοπικιλότητα. Αλλά παρόλα αυτά, όταν αναλύουμε ζητήματα βιοπικιλότητας, ενδεχομένως να υπάρχουν ακόμα τοξικές ουσίες στο, στα ύδατα. Και αυτό προφανώς ε, μας οδηγεί στο θέμα των διαταρακτών, στο θέμα των ορμονών. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Θα πρέπει όλες ε, αυτές οι μελέτες που πραγματεύονται ζητήματα τοξικολογίας να μάλλον όλες οι εκθέσεις που πραγματεύονται ζητήματα υδάτων να εξετάζουν και το θέμα των τοξικών ουσιών, οι οποίες μπορεί να έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες για όλα τα είδη και προφανώς και για τον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πόρτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ μου δίνετε το λόγο. Μια μικρή ερώτηση. Τι μέτρα σκοπεύει να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπιστεί το θέμα των λιμάτων από τα εργοστάσια επεξεργασίας λιμάτων. γιατί σε πολλές περιπτώσεις ε, δεν ξέρουν ε, τα κράτη-μέλη τι να κάνουν με τη λιματολάσπη αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος και εγώ να προσθέσω μια δική μου ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Τα κράτη-μέλη τα οποία εστερούν, που έχουν μείνει πίσω, τι θα πρέπει να κάνουν για να α, πληρούν τελικά τις πιο σημαντικές παραμέτρους όπως ορίζονται στην οδηγία για την επεξεργασία αστικών λιμάτων. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει επακριβώ τι θα πρέπει να γίνει. Ποια θα είναι τα πρώτα βήματα. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις λοιπόν, ο κ. Μαλγκάη για να απαντήσει. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ για τις ε, πολύ ουσιώδεις ερωτήσεις. Θα τις ομαδοποιήσω καταρχήν. Πρόεδρε, ως προς τη σημασία αυτού του θέματος για την κοινή γνώμη και για την κοινοποίηση προς το κοινό, με συνέπεια έχετε δίκιο. Γιατί δυστυχώς οι κύκλη ενημέρωσης είναι απότοκοι ενός μέσου που διανύει μία δεκαετία, την πρώτη δεκαετία. Γι' αυτό θα πρέπει να το εντάξουμε στα πλαίσια της επεξεργασίας ε, υδατολιμάτων γενικότερα. Και θα δείτε επιπτώσεις αυτής της οδηγίας και σε θέματα τοξικολογίας, γιατί τα αστικά ε, υδατολίματα είναι ένα μέσο που είναι πραγματικά συνεκτικό και συνεπές έτσι ώστε να υπάρχει πραγματική επεξεργασία ύδατος. Και αυτό ε, οδήγησε και σε μία οδηγία πλαίσιο για την επεξεργασία των υδάτων. Άρα χρειαζόμαστε μία ε, ολιστική προσέγγιση, να δούμε ποιοι είναι και οι επιμολυντές που θα πρέπει να απασχολήσουν τα κράτη-μέλη για να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το μέσο που είναι στο τέλος της πορείας, αλλά παράλληλα και την ποιότητα των ε, υδάτων των ποταμών, δηλαδή και μέτρα πέραν αυτού του απλού μέσου. Είπα ότι γι' αυτό το λόγο θέλουμε να προβούμε σε μία ενδελεχή αποτίμηση, δηλαδή πόσο συνεισφέρει αυτή η οδηγία ε, σε σχέση με τις τελικές επιπτώσεις. Και εδώ θα επανέλθω στα δύο ερωτήματα σε σχέση με τα φαρμακευτικά ε, λύματα και την τοξικολογία. Θα θέλαμε να δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει ε, από τις μονάδες επεξεργασίας λιμάτων. Είδαμε όμως ότι η απάντηση αυτή αφορά μία αδρή χρηματοδότηση και επενδύσει και το ζήτημα είναι ποιος θα καταβάλει το αντίτιμο. Εκείνοι που χρησιμοποιούν ε, τα αστικά λίματα ή εκείνοι που αγοράζουν τα φάρμακα και εδώ μιλάμε για την επεκτηνόμενη ευθύνη του παραγωγού σε σχέση με την φαρμακευτική στρατηγική που επεξεργάζεται η Επιτροπή. Το 2013 αναλάβαμε μία ε, δέσμευση ε, με βάση αυτό το προσχέδιο για τα ύδατα της Ευρώπης και ελπίζω αυτό το έγγραφο να εγκριθεί για να δούμε τι συμβαίνει και με τα φαρμακευτικά υπολείμματα στον υδάτινο όγκο και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα υπολείμματα. Ε, ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιούνται λιγότερο επιβλαβείς ε, ουσίες και φυσικά να δούμε ποιος θα καταβάλει το αντίτιμο, ο τελικός χρήση, χρήστης του σκευάσματος ή όχι. Και επειδή διαγράφονται αυτές οι τάσεις, βλέπουμε ότι η χρήση φαρμάκων θα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο στην Ευρώπη. Αυτή είναι μία ομάδα ερωτήσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκείνους που μίλησαν για απτή βελτίωση, αλλά υπάρχουν και ζητήματα για το τι συμβαίνει με την υλή ε, με βάση συγκεκριμένες νομοθεσίες, διότι η υλή σε αυτή δεν πρέπει να πηγαίνει στις ε, χωματερές. Επίσης υπάρχει ένα ε, άλλο μέσο για τη χρήση της ηλίως, όπου προβάλλουμε ποιοτικά κριτήρια και γι' αυτό προσπαθούμε να δούμε πώς η ποιότητα της ηλίως είναι τέτοια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θρεπτική ουσία, γιατί για τα μικροπλαστικά βλέπουμε ότι η ηλίς ε, εμπεριέχει ορισμένες από τις ουσίες που είχαμε ε, δει εκ των προτέρων, άρα τίθεται και θέμα ασφάλειας των τροφίμων. Θα πρέπει να εργαστούμε περαιτέρω επί του θέματος, αλλά είναι περίπλοκο ως προς τις ε, παραβάσεις και για τα παλαιότερα κράτη-μέλη δυστυχώς υπάρχει μεγάλος αριθμός διαδικασιών επί παραβάση. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τις χώρες άμεσα, αλλά δυστυχώς πρέπει να προσφύγουμε σε ένδικα μέσα πολλές ε, φορές. Είναι πολύ δύσκολο να γίνεται διάλογος με κάθε περιφερειακή κυβέρνηση. Ελπίζω με αυτή τη συλλογική προσπάθεια να μπορέσουν οι περιφέρειες να αντιμετωπίσουν αυτή την ε, νομική πρόκληση. Και αυτό τώρα το συσχετίζω με την ε, ερώτηση της Προέδρου για το τι μελιγενέστε. Έχει μεγάλη σημασία το θέμα της διακυβέρνησης διότι πολλές φορές το θέμα των επενδύσεων προκύπτει όταν έχουμε να κάνουμε με μικρότερες ε, οντότητες ή κοινότητες που πρέπει να προβάλλουν ένα πρόγραμμα. Και ό,τι, όπως και να έχει, εμείς είμαστε ουδέτεροι, αλλά και η κεντρική κυβέρνηση θα πρέπει να βοηθήσει τις μικρές κοινότητες και παρόχους να συνεργαστούν. Όταν υπάρχει νομική παράβαση, επιμένουμε σε ένα ε, αξιόπιστο master plan για να ξέρει η κυβέρνηση τι χρειάζεται, πού χρειάζεται, ποια είναι η χρηματοδότηση, από πού προέρχονται ε, τα χρήματα, προέρχονται από δασμούς, από ευρωπαϊκούς πόρους και ούτω καθεξής. Πιστεύουμε ότι με αυτή τη στρατηγική προσέγγιση θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ελπίζω να απάντησα τις, ε, στις περισσότερες ερωτήσεις. Τώρα, ως προς τη συνοχή των, ε, της εργασίας των Επιτροπών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσπαθούμε να έχουμε μία συνεκτική προσέγγιση, αλλά πολλές φορές ε, δεν γνωρίζω πώς έχουν συγκεκριμένες επιμέρους ε, συζητήσεις. Αυτό όμως που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δούμε τι θα γίνει με την πρόταση για το πόσιμο νερό, γιατί για παράδειγμα για τα λοιπάσματα, εγώ δεν, δεν γνώριζα πώς είχε εξελιχθεί η συζήτηση. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις περιφέρειες στρατηγικά, δηλαδή το πόσιμο νερό να μην το δούμε στο τέλος αυτής της πορείας, αλλά οι περιφερειακές κυβερνήσεις να δούνε ποιοι είναι οι κίνδυνοι έτσι ώστε να έχουμε μια πιο συνεκτική προσέγγιση ε, υποστήριξης της γεωργίας σε συγκεκριμένες περιφέρειες όπου υπάρχει πρόβλημα του υδροφόρου ορίζοντα ή τι γίνεται με τους ε, βιομηχανικούς ε, ρήπους και εκπομπές. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ενδυνάμει πηγές ρήπανσης Εάν θέλετε μπορώ να επανέλθω αν υπάρχουν περαιτέρω ερωτήματα. Υπάρχει μία ερώτηση πράγματι. Κυρία Σχαϊοπύρικα, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξηγήσεις που μας έδωσε. Αλλά είπατε ότι σε ό,τι αφορά την λιματολάσπη, ότι μιλάμε για την, τον εμπλουτισμό και σε ό,τι χρήση τους όσοι λιπάσμα. Τι γίνεται όμως με τα λιπάσματα από τον αγροτικό τομέα και θα ήθελα να έχω μια γραπτή απάντηση γιατί θεωρώ ότι εδώ υπάρχει μεγάλο δυναμικό και θα ήθελα να σας πω ότι ενδεχομένως να καταθέσω και τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν απαραίτητο το λόγο για να απαντήσετε τώρα. Αν θέλετε να απαντήσω γραπτά για να μπορέσω να συμβουλευτώ και τους αρμόδιους συναδέλφους. Μάλιστα λοιπόν, λέει η Πρόεδρος. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε και η ανταλλαγή απόψεων για το, την ε, οδηγία για την επεξεργασία αστικών κολλημάτων. Σας ευχαριστώ και να περάσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Και πάλι ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ευρωπαϊκές δράσεις, για την βελτίωση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Ο κ. Ρόμπερτ Κόνραντ Γιούνετ, διευθυντή επικεφαλή τη Γενική Διεύθυνση Environment, έχει το λόγο. Α πάρετε πρώτο το λόγο λοιπόν εσεί και μετά στη διαδικασία κάτσου θα πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι. Ο κ. Κόνραντ έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ και για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε το σχέδιο δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, περιβαλλοντική συμμόρφωση και διακυβέρνηση που εγκρίθηκε στι 18 Ιανουαρίου. Για να δω πώ μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Μιλάμε λοιπόν για ένα πακέτο το οποίο εγκρίθηκε τον Ιανουάριο Έχουμε την ανακοίνωση, το έγγραφο εργασία και την απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δημιουργία μια νέα ομάδα εμπειρογνωμόνων. Η βασική, αν θέλετε, λογική της, ε, των πακέτων ε, περιβαλλοντική συμμόρφωση είναι η εξή. Μετά από πολλά χρόνια εμπειρία με θέματα ελλειπούς εφαρμογής και χρησιμοποιώντας ε, και το έργο του ακαδημαϊκού κλάδου και του ίδιου του κλάδου στον τομέα αυτό, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι για να λειτουργεί η περιβαλλοντική συμμόρφωση χρειάζονται τρία βασικά στοιχεία, τρει βασικοί πυλώνες. Καταρχά προώθηση της συμμόρφωση που σε ό,τι αφορά δηλαδή δράσεις και ενέργειε, όσο που είναι ενημέρωση, πληροφόρηση, διαφάνεια, χορήγηση χρηματοδότησης. Ύστερα έχουμε τις επιθεωρήσεις και του ελέγχου και τέλο, εξίσου σημαντικό πυλώνα το στοιχείο της ε, υλοποίηση, τη εφαρμογή. Και προκειμένου να σα εξηγήσουμε όλους αυτούς τους τύπους συμπεριφοράς, να σα πούμε το εξή ότι οι δικαιούχοι ε, έχουν πολύ μεγάλη γκάμα σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση. Έχουμε τους πρωταθλητές, έχουμε και τους εγκληματίες. Και φυσικά οι διάφορες, ε, οι διάφοροι τύποι αντίδρασης ε, προσαρμόζονται στους τύπους αυτούς. Ε, έχουμε λοιπόν την επιβράβευση, έχουμε την χρηματοδότηση, την κατάρτιση, τους ελέγχους, την εφαρμογική υλοποίηση ως αντιδράσεις. Στο πακέτο λοιπόν προσπαθούμε να καταγράψουμε την πλήρη γάμα αντιδράσεων, προκειμένου να καταλήγουμε σε κάθε περίπτωση στην πλέον κατάλληλη αντιδράση. Αντιλαμβανόμαστε και υπάρχουν και σωστή τεκμηρίωση σε ό,τι αφορά και τη σχετική αξιολόγηση περιβαλλοντικής συμμόρφωσης. Οι μηχανισμοί λοιπόν συμμόρφωσης αποτελούν όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα, μία από τις βασικές αιτίες ελλειπούς εφαρμογής του κινητικού κεκτημένου στα κράτη-μέλη. Η εφαρμογή λοιπόν και η υλοποίηση δεν συζητιέται συνήθως με συνδυασμένο τρόπο. Και έτσι λοιπόν υπήρχε η αξίωση να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα υψηλού επίπεδου η οποία θα επέτρεπε ανταλλαγή των επιρρογνωμόνων για τέτοια ζητήματα εξασφάλισης συμμόρφωσης. Επίσης, τονίζεται η ανάγκη συνεργασία των εμπειρογνωμών από διάφορου κλάδου. Να σα ε, διαβεβαιώσω ότι όταν μιλάμε για εμπειρογνώμονε, μιλάμε για του επιθεωρητέ σε ό,τι αφορά την πρακτική επιτόπου. Μιλάμε δηλαδή για τους επιθεωρητές των ε, εργοστασίων, των εγκαταστάσεων, των ε, πράσινων εγκαταστάσεων που αντιμετωπίζουν και ασχολούνται με διάφορους κλάδους συμμόρφωση για το περιβάλλον. Μιλάμε επίση για του εισαγγελεί, για τι αστυνομικέ δυνάμεις και για το δικαστικό σώμα. Όλοι αυτοί λοιπόν οι εμπλεκόμενοι φορεί, τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι οι επιρρογνώμονε με του οποίου έχουμε συνεργαστεί μέσα από διάφορα δίκτυα επί σειρά ετών και όλοι αυτοί λοιπόν θα πρέπει να εμπλακούν στην παρούσα φάση σε επίπεδο κρατών μελών αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων προκειμένου να σχηματιστεί αυτή η πλατφόρμα που θα μας δώσει την δυνατότητα να συνεργαστούμε πραγματικά, να ανταλλάξουμε απόψεις με συστηματικό και διαθρώμενο τρόπο. Κάτι άλλο. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η πληροφόρηση γίνεται από κάτω προς τα πάνω και αυτό προφανώς δεν είναι ο βέλτιστος τρόπος. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη καθοδήγηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα για κάποιου τομεί. Και φυσικά υπάρχουν και πρακτικέ προκλήσει, οι οποίε εμφανίζονται σε όλη τα επίπεδα, σε επίπεδο κρατών μελών και για τους επιθεωρητές και για τους δικαστές και για όλα τα διάμεσα τους ενδιάμεσους κλάδους. Τέλος, η εξασφάλιση συμμόρφωσης προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και διαπιστώνουμε όλο και πιο πολλές νέες τεχνολογίες οι οποίες καθορίζουν την αποτυχία, την επιτυχία της παρατήρησης, ε, της χορήγησης και διανομής δεδομένων μέσω διαδικτύου, μέσω ε, εφαρμογών, μέσω άλλων συστημάτων φιλικών ή μη προς το χρήστη. Το αποτέλεσμα λοιπόν, το πόρισμα της έρευνα σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τις δράσεις οι οποίες α, προτείνεται στο σχέδιο δράσης. Εννέα στον αριθμό τέτοιες δράσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι στο γράφημα υπάρχει μια, γίνεται μια απόπειρα να δώσουμε μια απάντηση στις βασικές αυτές προκλήσεις. Ας ξεκινήσουμε από την δεξιά πανογωνία. Ανάπτυξη συστήματων δορυφορικών για να υπάρχει η καλύτερη αξιοποίηση των εθνικών συστημάτων για την παρατηρήση και παρακολούθηση της Αίγης. Συνεργαζόμαστε στο πρόγραμμα Κοπέρνικος και είναι μία πρόκληση το πρόγραμμα αυτό, το Κοπέρνικος, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη και πιο συστηματική εξασφάλιση της συμμορφώσης. Επίσης, θέλουμε να δώσουμε στα κρατημέλη καλύτερο feedback για την απόδοσή τους. Να αναπτύξουμε ένα πλαίσιο αξιολόγησης, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει κάποιους δείκτες βασικούς για την απόδοση, το οποίο θα αξιολογεί λοιπόν τα κρατημέλη. Προσπαθούμε να δίνουμε καλύτερη καθοδήγηση. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση στην Ήπετρο. Ένα έγγραφο καθοδήγησης με τις βελτιστές πρακτικές σε ό,τι αφορά την Ήπετρο, σε ό,τι αφορά τα θέματα ύδατος και φωτός. Επίσης, θέλουμε να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση κατά των ε, απορριμμάτων και των εγκλημάτων κατά της ε, αγριάς ζωής. Να επικεντρωθούμε λοιπόν στο θέμα αυτό. Φυσικά η ενημέρωση, η πληροφόρηση, η δυναμή της γνώσης αν θέλετε και των δεδομένων των βελτιστών πρακτικών, τα υλικά αναφοράς ε, και η προώθηση των διαφόρων δυνατότητων χρηματοδότησης σε τέτοια ζητήματα. Και η σύσταση ενός κόμβου, αν θέλετε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περαιτέρω. Προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης. Εδώ πολλά ενδιαφερόμενα μέρη μας δήλωσαν ότι θα πρέπει να εντοπιστούν οι επαγγελματικές δεξιότητες που χρειάζονται για τους επιθεωρητές και να προωθηθούν μέσα από προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης για να προωθηθεί η αριστεία σε αυτό το επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Και φυσικό θέλουμε να βοηθήσουμε και τους επιθερωτές και τις ε, αρχές εφαρμογής του νόμου προκειμένου να συνδυάσουν τις ε, ικανότητές τους και τις δυνάμεις τους για την ε, αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω, για παράδειγμα, αξιολογήσεων από ομοτήμους, κοινών προγράμματων κτλ. Έχουμε επίσης ε, τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την επιθεώρηση των ε, εργοστασίων επεξεργασίας λιμάτων και τέλος ένα βασικό στοιχείο είναι να υπάρχει η δυνατότητα για τους πολίτες και για τις ΜΚΟ, για τους τοπικούς φορείς, να υποβάλουν καταγγελίες αν κάτι θεωρούν ότι δεν πάει καλά. Τεκμηρίωση λοιπόν των βέλτιστων πρακτικών και αντιμετώπιση καταγγελιών για ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον σε επίπεδο κρατών μελών και συνεργασία μεταξύ κρατών μελών για την διανομή των βέλτιστων αυτών πρακτικών. Αυτές λοιπόν είναι οι εννέα δράσεις οι οποίες θα εφαρμοστούν το 2018-2019. Επίσης, ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα μια νέα ομάδα, επίσημη ομάδα υψηλού επίπεδου που συμπεριλαμβάνει τους εμπειρογνώμονες και χαρήκαμε που διαπιστώσαμε ότι τα κράτη-μέλη αντιμετώπισαν με σοβαρότητα την πρόκληση αυτή και ήταν πολύ καλή η συμμετοχή και από τις εθνικές κυβερνήσεις, από τα Υπουργεία, αλλά και από τις εθνικές αρχές επιθεώρησης. Και προφανώς Προσκαλέσαμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και άλλα ευρωπαϊκά όργανα και υπηρεσίε στην ε, πρώτη μας συνάντηση που θα καθορίσει και το πρόγραμμα ή στη δεύτερη ενδεχομένως το Δεκέμβριο θα καθοριστεί πιο επισταμένο στο πρόγραμμα. Βλέπετε λοιπόν ένα χαρτί ο οποίο περιλαμβάνει τι ε, δομέ διακυβέρνηση και τι διάφορε οργανώσει. Βλέπετε λοιπόν τα κράτη-μέλη τα οποία συνεργάζονται με τα περιβαλλοντικά δίκτυα, τα οποία έχουν ρόλο κλειδί, γιατί αυτά κάνουν ουσιαστική, ουσιαστικά τη δουλειά. Αυτά μα δίνουν τα δεδομένα που χρειαζόμαστε. Θέλουμε λοιπόν να σχηματιστούν και ομάδε εργασία και workshops, εργαστηρία προκειμένου να είναι στοχευμένη η ανταλλαγή απόψεων σε υψηλό επίπεδο για όλα τα ζητήματα διακυβέρνηση. Και εδώ τα όσα συμφωνήθηκαν στο άρχους. Και φυσικά θα υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ομάδων εργασία σε ό,τι αφορά τους διάφορες ενότητες ε, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το νερό, τη φύση και το καθεξής. Αυτά είχα να σας πω. εισαγωγικά αυτές ήταν οι διάφορες γραμμές. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay, thank you very much for the presentation. Now, colleagues would like to... Συνάδελφοι, ποιος θα ήθελε να λάβει το λόγο σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Η κυρία Πέρικ. Πρόεδρε, άλλη μια καλή παρουσίαση. Εγώ θα ήθελα όμως να ξαναθέσω την ερώτηση που έθεσα και προηγουμένως. Όλα καλά και όλα ωραία. Αλλά όταν μιλάμε για την μη επεξεργασία των λιμάτων, αυτό έχει επιπτώσεις και για τα κανάλια και για τους ε, ποταμούς. Και δεν έχουμε στοιχεία, γιατί τα στοιχεία που μας στέλνουν τα Συμβούλια ε, επεξεργασία ε, των Υδάτων είναι ανησυχητικά. Και ποιες είναι οι συνέπειες αυτές και για τον κόσμο που ζει στην Ήπεθρο. Ευχαριστούμε κάποιος άλλος. Η κυρία Γκροστέτ. Εγώ θα θα μιλήσω για το νερό αλλά τον αέρα. Τέλη Ιανουαρίου η Επιτροπή συγκάλεσε νέα κράτη μεταξύ των οποίων και τη Γαλλία για μία ε, συνάντηση της τελευταίας ευκαιρίας και οι χώρες αυτές ε, είχαν 10 μέρες για να υποβάλουν ένα αξιόπιστο σχέδιο έτσι ώστε να ε, εξαλειφθεί το διοξίδιο του αζότου στον αέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο τα εξώδικα αρκούν, γιατί όταν ε, ε, λέμε σε κράτη-μέλη έχετε 10 μέρες για αξιόπιστες δράσεις, αυτό δεν είναι απλό. Θα ήθελα όμως να μου πείτε αν είναι δυνατόν και σήμερα που έχουμε φτάσει. Ο κύριος Φλόρενς. Θα μπορούσα να βάλω ένα δίσκο τον οποίο τον έχουμε ακούσει και πριν από 20 χρόνια. Με μεγάλη χαρά ακούω τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις προθέσεις της για να βελτιώσει στο μέλλον ορισμένα πράγματα ή εν πάση περιπτώσει σε όσα δεν, έχει, δεν έχουν κάνει τα κράτη-μέλη. Ξέρετε, εγώ συμμετείχα και έγραψα τότε το 1994 την ε, οδηγία άμα, για τα ύδατα. Και ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί αυτή η οδηγία, ξέρετε, στην χώρα μου. Αν είχα κάνει τα μαθήματά μου στο σχολείο τόσο άσχημα όσο κάνει η χώρα μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έμεινα μεταξαστέως. Μα γιατί αφήνετε τέτοια μεγάλα κενά. Υπάρχουν κρατήδια στη Γερμανία που τα παραμποδίζουν όλα αυτά και μου κάνει εντύπωση το γεγονό ότι τα ανέχονται αμα, αυτά οι επίτροποι στους Ολλανδούς τους α, ε, τιμώρησαν αυστηρά και είναι αυστηροί με αυτού. Άλλο του αφήνουμε, ξέφραγο αμπέλι. Προσέξτε λοιπόν, όλα αυτά που να μου νομοθετείτε να υλοποιούνται κιόλα. Μπορεί κάποια πρότυπα να μην είναι τόσο ιδανικά ή εν πάση περιπτώσει να μην ανταποκρίνονται στι προσδοκίε ε, κάποιων ευρωβουλευτών. Αλλά το γεγονό ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν εφαρμόζουν επί σειρά ετών τέτοιε αποφάσει με αφήνει έκπληκτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξίζει να ονομάζεται Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είσαστε υποτίθεται θεματοφύλακα των Συνδικών. Και μερικά πράγματα μπορεί να μην αρέσουν σε κάποιου, αλλά αυτό που διαπιστώνω είναι ότι στου Ολλανδού συναδέλφου θέτεται πάρα πολλέ αυτέ τι προδιαγραφέ και υπάρχουν άτομα στο νότο τη χώρα μου που δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση. Είναι πραγματικά αδιανόητα αυτά. Απευθύνω λοιπόν έκκληση, θερμή έκκληση για τα τελευταία αυτά χρόνια. Ας εφαρμοστούν επιτέλους αυτές οι προδιαγραφές. Yes, thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος άλλος. Θα ήθελα και εγώ να υποβάλω μία δική μου ερώτηση. Το αντιμετωπίζετε χώρα προς χώρα το θέμα σε σχέση με την βελτίωση της διακυβέρνησης, γιατί όπως φάνηκε από την προηγουμένη συζήτηση πολλές φορές η εφαρμογή, η εφαρμογή δεν μπορεί να γίνει γιατί υπάρχει έλλειψη διακυβέρνησης. Τώρα το λόγο έχει και πάλι η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Φοβάμαι ότι δεν είμαι σε θέση να απαντήσω τις συγκεκριμένες ερωτήσεις για τα ύδατα και τον αέρα, όμως θα προσπαθήσω να απαντήσω για τη διαδικασία διακυβέρνησης με βάση το πρόγραμμα δράσης. Ένα από τα πράγματα που αναπτύσσονται τώρα είναι ένα πλαίσιο αξιολόγησης. Όπως γνωρίζετε, είχαμε την πρώτη αναθεώρηση του περιβάλλοντος όπου υπάρχουν οι πρώτοι δείκτες διακυβέρνησης και τώρα θα επεκτείνουμε και θα καταρτήσουμε περαιτέρω τους δείκτες αυτούς έτσι ώστε να επεκτείνουμε και το κεφάλαιο 5 ακριβώς για να έχουμε πιο, μια πιο ολιστική εικόνα της κατάστασης της διακυβέρνησης στα κράτη-μέλη. Αυτό παρουσιάστηκε και στη συνάντηση των κρατών σε αυτό το φόρουμ και γι' αυτό πιστεύουμε ότι σε αυτή την ε, κοινή προσπάθεια θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μία πληρέστερη εικόνα το 2019 για το πώς λειτουργεί δηλαδή στα κράτη-μέλη. Είναι μία διαδικασία που έχει ξεκινήσει και θα βελτιωθεί όσο προχωρούμε. Ελπίζουμε όμως να έχουμε μία πιο εμπεριστατωμένη γνώμη για τις χώρες καθεαυτές, καθώς και την ε, διακυβέρνηση σε όλα τα κράτη-μέλη. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ. Ως προς τα... το... το νερό και τον αέρα, μπορείτε να περάσετε τα ερωτήματα στους συναδέλφους έτσι ώστε να λάβουμε μια απάντηση από την Επιτροπή. Άρα λίγη και η συζήτηση σε αυτό το θέμα και περνάμε στο επόμενο Again, an exchange of views. Ανταλλαγή απόψεων για την ενδιάμεση αναθεώρηση και το μέλλον του προγράμματος για την υγεία. Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε τον κύριο Ιορδάνου, Διευθυντή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να σας δώσω κάποιες προφορές για την αξιολόγηση και μετά να μιλήσω για τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον. Παρουσιάσαμε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στις 11 του περασμένου Οκτωβρίου την έκθεση αξιολόγησής μας που βασίζεται στα ευρήματα αλλά και στις συστάσεις που ε, υπάρχουν σε μια εξωτερική μελέτη που εκποδήθηκε από το Μάιο του 16 μέχρι το Μάιο του 17 και τα πορίσματα της μελέτης αυτής της εξωτερικής αξιοποιούνται για τη βελτίωση της εφαρμογής του προγράμματος για την υγεία την περίοδο 18 με 20 και θα είναι και χρήσιμα για την ε, περίοδο μετά το 20. Το τρίτο πρόγραμμα για την υγεία είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο για το συντονισμό πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να συμπληρώσει ε, να στηρίξει και να προσθέσει αξία στις προσπάθειες των κρατών μελών για να βελτιώσουν την υγεία των πολιτών τους και να μειωθούν οι ανισότητες. Η συγκεκριμένη στόχη είναι να προαχθεί η υγεία, να προστατευτούν οι Ευρωπαίοι από σοβαρές διασυνοριακές απειλές υγείας, να συμβάλλει σε αποτελεσματικά και βιώσιμα συστήματα υγείας, να ε, βελτιώσει την πρόσβαση σε καλύτερη περίθαλψη και καλύτερο σύστημα υγείας. Επομένως, η ενδιάμεση αξιολόγηση τα τρία πρώτα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος. Έγινε πολύ νωρί για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ποσοτικά κατά πόσο θα πετύχουμε τους στόχους του προγράμματος, γιατί οι περισσότερες δράσεις εκτείνονται πέρα από την τριετή περίοδο της ενδιάμεσης αξιολόγησης και ε, τα, τα τελικά αποτελέσματα των δράσεων του 2015 θα είναι ε, διαθέσιμα στα τέλη του 2018. Έχουμε μεγάλα επιτεύγματα. Έχουμε 24 ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς για σπάνιες ασθένειες προς το παρόν. Αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα. Στηρίζουμε τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τη δυνατότητά τους να ανθίστανται και να ε, ανταπεξέρχονται σε επιδημίες, όπως ο ιός έμπολα, όπως ε, ο ιός ζήκα και συμβάλλουμε την, στην μεταναστευτική πολιτική γιατί συμβουλεύουμε τα κράτη-μέλη πώς θα ανταποκριθούν στις ανάγκες υγεία των προσφύγων και μεταναστών και προσφέρουμε κατάρτιση μέσω του προγράμματος, ανταλλάσσονται οι καλές πρακτικές και σε τομείς όπως ε, ο έγκυρος έλεγχος για το καρκίνο, για το νιό HIV, για την πρόληψη από τη φυματίωση, ε, ε, για την μείωση της κατανάλωσης των πνευματοδών ποτών. Για, επίσης έχουμε ενίσχυση της ηλεκτρονικής υγείας, των ηλεκτρονικών εφαρμογών στον τομέα της υγείας. Συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Εθνικά Συστήματα Υγείας και Πολιτικές, αλλά και με τον ΟΣΑ για να έχουμε σειρά εκθέσεων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο 28 κρατών μελών. Αυτά δημοσιεύθηκαν τον Νοέμβριο του 16 και του 17. Ετήσια δημοσίευση δηλαδή. Επίσης να σας πω ότι μετά από αυτή την αξιολόγηση Υιοθετήσαμε μέτρα απλούστευσης για να μπορέσουν οι φορείς να υποβάλουν προτάσεις και να διαχειρίζονται τις ενισχύσεις ηλεκτρονικά. Απλουστεύσαμε τους κανονισμούς για τη χρηματοδότηση και τον τρόπο αξιολόγησης. Έχουμε πιο στρατηγική άποψη για την ενδιάμωση αξιολόγηση και τις ενδιάμεσες προοπτικές πρέπει να είναι ένα ευέλικτο εργαλείο χρηματοδότησης που να καλύπτει απρόβλεπτες ανάγκες, όπως ήταν η κρίση με τον ιό έμπολα ή οι ανάγκες σε υγεία και σε περίθεψη των προσφύγων και μεταναστών που ήταν ε, κάτι ε, το έκτακτο και όχι το προβλεφθέν. Στόχος μας είναι να ε, πετύχουμε προστιθέμενη αξία, να έχουμε σημαντικά αποτελέσματα και να τα αναδείξουμε, να σηκώσουμε αυτό το θέμα ψηλά, και η έκθεση αξιολόγησης βασίζεται στις υπηρεσίες που δίδονται ε, στους αξιωματικούς συνδέσμους για το πρόγραμμα και στα κράτη-μέλη. Ξεκινήσαμε και δημόσια διαβούλευση και είχαμε 130 συνεισφορές. Ευρεία η στήριξη για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής δράσης στον τομέα της υγείας, το 97% των απαντώντων Συμφώνησα στο ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία σε θέματα υγείας είναι απαραίτητη και θα πρέπει να διατηρηθεί. Δύο λόγια για το μελλοντικό προγραμματισμό και τις προοπτικές μας με τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος. Αυτή τη στιγμή συζητούμε πώς θα διαμορφώσουμε με τον καλύτερο τρόπο νέο πρόγραμμα και νέο, νέους χρηματοοικονομικούς θεσμούς, χρηματοδοτικούς θεσμούς, για να είναι πιο ευέλικτοι αυτοί, να έχουν καλύτερη συνέργεια, να είναι πιο αποτελεσματικοί. Οι μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα της υγείας πρέπει να είναι πιο στοχευμένες, γιατί ο προπολογισμό είναι περιορισμένος. Πρέπει να ενισχυθούν οι δράσεις που θα κομίσουν τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία. Να προτεραιότητα είναι να επιλεγούν τα κατάλληλα προγράμματα έτσι ώστε τα εθνικά συστήματα υγείας να επενδύσουν έξυπνα στην υγεία, στην καινοτομία και στην έρευνα. βλέπουμε πώς μπορεί να έχουμε αποτελέσματα εάν συνεργαστεί αυτό το χρηματοδοτικό μέσο με άλλα ε, χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προωθώντας την ευρύτερη ε, ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκοστέτ. έχει το λόγο για το υφιστάμενο πρόγραμμα για την υγεία. Είστε εισηγήτρια στη σχετική έκθεση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι αληθές ότι αυτό το τρίτο πρόγραμμα για την υγεία με πρικοδότηση 500 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να φαίνεται ψίχουλα. Ψίχουλα είναι αυτά για να μειωθούν οι ανισότητες στις πολιτικές υγείας στα 27 κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά, είναι χρήσιμο, γιατί στηρίζει τους στόχους μας για την υγεία. Επομένως, νομίζω ότι καταρχάς πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, να μην κάνουμε δύο φορές την ίδια δουλειά. Και δεν είμαι σίγουρη ότι δεν γίνεται αυτό. Θα έπρεπε να έχει λυθεί αυτό το θέμα και δεν έχει λυθεί. Να καλύψουμε τα κενά. Υπάρχει πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας και εν μέρη θα χρηματοδοτεί τη σχετική επιτροπή από το πρόγραμμα για την υγεία. Για να είναι αποτελεσματική αυτή η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών πρέπει να τις δώσουμε τους απαραίτητους πόρους. Άρα μας λέτε για περιορισμού στον προϋπολογισμό. Μας ανησυχεί αυτό, τα μάλα. Και ε, έμαθα ότι για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έμαθα ποιες είναι οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κοιτάξτε, εγώ νόμιζα ότι το πρόγραμμα για την υγεία μπορεί να γίνει τελικά υποκατηγορία ενός ευρύτερου προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά» με αναφορά διατροφική ασφάλεια, υγεία των ανθρώπων, υγεία των ζώων και ε, υγεία των φυτών. Κοιτάξτε, δεν έχω πρόβλημα να συνδέσουμε την υγεία με την ανάπτυξη. Και τότε το, το τρίτο πρόγραμμα έτσι έπρεπε να είχε ονομαστεί. Πρόγραμμα για την υγεία, για την ανάπτυξη. Όμως είμαι κάθετα αντίθετη σε οποιαδήποτε στρατηγική. Τελικά καταλήξει να κάνει το πρόγραμμα της υγείας να έχει δεύτερο αγωνιστικό ρόλο και όχι πρωταγωνιστικό, να γίνει απολύτω δυσνόητο και ακατανόητο για τους πολίτε μα. Η υγεία είναι κάτι που αφορά καθημερινά στην καθημερινότητα όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και το, η ενιαία αγορά του είναι πολύ λιγότερο εύγλωτη σαν έννοια. Ε, δεν μιλάει τόσο καλά, δεν απευθύνεται τόσο καλά στον Ευρωπαίο πολίτη. Και άλλωστε δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα στο ίδιο καλάθι. Την υγεία των ζώων, την καλή διαβίωση των ζώων, την ε, ευημερία αν θέλετε ή την ε, υγεία των φυτών. Μπορούμε να μιλούμε για κάτι τέτοιο να το βάζουμε στο ίδιο καλάθι με την υγεία των ανθρώπων. Σε κάθε περίπτωση, οι προτάσει σα για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο νόμιζα ότι ήταν σύμφωνε με τι δικέ μα. Εγώ ζητώ από όλου του συναδέλφου που ανησυχούν για τα θέματα της υγείας των ανθρώπων, που είναι πραγματικά ένας τομέας που μπορούμε να αποδείξουμε την αξία ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής ένα χρόνο από τις ευρωεκλογέ, είναι ε, ε, σημαντικό να τους δείχνουμε ότι δεν ε, παραμελούμε αυτά τα θέματα. Εγώ θα δώσω τη μάχη για να τα καταφέρουμε, αλλά βασίζομαι στους συναδέλφους από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσο πιο πολλοί άριθμοι είμαστε, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ, η Συμπρόεδρη της ομάδα Εργασίας ε, για την Υγεία και το Περιβάλλον. Η κυρία Καβεσόν Ρουίς. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Γκροστέτ. Είμαι ιδιαίτερα ανήσυχη γιατί όπως ε, προελέχθη υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Θα αποτελέσει μέρος αυτό το πρόγραμμα ενός μεγαλύτερου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι θα εξαφανιστεί. Αυτό το ακούσαμε μόνο, αλλά το αφήνω, γιατί ακόμα και η Γενική Διεύθυνση Υγείας φαίνεται ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσει να υπάρχει. Αυτό με απασχολεί γιατί τα θέματα υγείας είναι πολύ σημαντικά και έχουν προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο φυσικά. Υπάρχει θέμα εθνικών υποχρεώσεων, αλλά και η ευρωπαϊκή νομοθεσία μας επιβάλλει να έχουμε υψηλές προδιαγραφές υγείας σε όλους τους τομείς. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε το πλαίσιο υγείας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο απολογισμός που προβάλλεται βγαίνει από αυτό το πρόγραμμα και το ζήτημα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, προκλήσεις γιατί νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να υπάρξει ε, χρηματοδότηση από αυτό το πρόγραμμα και μέσα στα πλαίσια του πολιετούς ε, δημοσίου πλαισίου. Και γι' αυτό τελικά έχουμε μεγάλη ανησυχία γιατί τα προγράμματα με τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τους πολίτες και για την οικονομία φαίνεται ότι εξαφανίζονται. Και στο πολιετές την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια ψηφίσαμε το πιδελταπί, αλλά δεν έγινε λόγος για προγράμματα υγείας, το οποίο σημαίνει ότι μάλλον θα εξαλειφθεί. Και σε αυτό αντιτασσόμαστε στεναρά. Ο κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συμφωνώ με όσα προελέχθησαν σήμερα Νομίζω ότι δεν θα ήταν ε, σωστό η υγεία να είναι κάτι το συμπληρωματικό σε άλλους τομείς. Αν δείτε τις τάσεις που διαγράφονται στον τομέα υγείας, θα πρέπει η υγεία να είναι στην εμπροστοφυλακή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολίτες σαν και εμένα κατανοούν ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ε, προσθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερη προσθέμενη αξία χωρίς να τροποποιήσουμε τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Με την ε, πείρα μας και την πραγματογνωμοσύνη μπορούμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα. Συμφωνώ με την κυρία Γκροστέτ ότι αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να συνεχιστεί. Έχω και ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια είναι η ανταπόκριση των ε, κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι τα κράτη-μέλη θα κάνουν πολύ περισσότερα, αλλά υπάρχει διαφορά στην προσέγγιση των κρατών μελών. Ξέρουμε ότι η Επιτροπή ε, προέβαλε πολλά επιχειρήματα, αλλά πώς ανταποκρίθηκαν τα κράτη-μέλη στην προσφορά της Επιτροπής. Κύριε Φράι Πέρεκ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η κυρία Γκροστέτ νομίζω ότι μίλησε με ξεκάθαρα λόγια μιλάμε για την ενιαία αγορά, αλλά εδώ μιλάμε για τον άνθρωπο. Μιλάμε για τα μωρά, για τους νέους, για τους ε, ηλικιωμένους, για όλα τα άτομα. Μιλάμε για όλα αυτά τα άτομα και όλα αυτά έχουν και οικονομικές επιπτώσεις. Συμφωνούμε μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου, αλλά αποφεύγουμε την ουσία του ζητήματος. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα και εγώ από πλευρά μου να ξέρω πώς θα αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά, πώς θα πει στο επίκεντρο και μια άλλη προοπτική. Στην ε, Ολλανδία, για παράδειγμα, το θέμα των φαρμακείων, των φαρμάκων και έρχεται ε, ο κόσμος και μας ρωτάει, μα τι κάνετε στην Ευρώπη. Τα βάζουμε όλα αυτά στο ίδιο καλάθι με τα υπόλοιπα. Και θεωρώ ότι αυτό δεν μπορεί να είναι η στάση της Επιτροπής μας, ούτε και του Συνολικού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ο κ. Ζωρίνιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πέρσι το Μάιο υπέβαλα ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν υπάρχει επαρκής ε, εναρμόνιση στις πρακτικές εμβολιασμού στα κράτη-μέλη και ρώτησα την Επιτροπή τι προτίθεται να κάνει για να προβάλλει αυτή την εναρμόνιση γιατί είναι πρωταρχικό μέλημα κάθε κράτους μέλους. Για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την ε, εναρμόνιση ως προς τα προγράμματα εμβολιασμού, γιατί σε ορισμένα κράτη-μέλη είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, σε άλλα όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση από κράτος σε κράτος, αλλά μου ανέφερε ότι στο πρόγραμμα αυτό υγείας θα υπάρξει κοινή δράση που θα συγχρηματοδοτηθεί για αυτές τις πρακτικές εμβολιασμού. Αυτό το θέμα ε, είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μου, διότι υπάρχουν πολύ μεγάλα κρούσματα ηλαράς, τα οποία πρέπει να ε, αντιμετωπιστούν. Θα πρέπει να υπάρχει μία καλύτερη διαπαιδαγώγηση σε θέματα εμβολιασμού, έτσι ώστε να προλαμβάνονται ασθένειες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κάποιος άλλος. Εάν όχι, ο κύριος Ράιαν έχει και πάλι το λόγο για να σχολιάσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως προς τα θέματα που εφήγησαν, καταρχήν τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς έχουν κινήσει την εργασία τους και προσπαθούμε να τα επεκτείνουμε. Δεν θέλουμε να επεκτείνουμε τα δίκτυα πάρα πολύ έως ότου τα 24 αρχικά δίκτυα μπορέσουν να λειτουργήσουν έμπρακτα. Ε, και γι' αυτό ζητούμε και τα διάφορα, ε, τη συνδρομή των, ε, της πληροφορίας και των ε, τεχνολογιών, των νέων τεχνολογιών και θέλουμε να δούμε κατά πόσο μπορούν να επεκταθούν βάσιμα. Πολύ αναφερθήκατε στην ε, τεχνολογική αξιολόγηση που θα αποτελέσει αντικείμενο μιας νομοθετικής ε, πρότασης, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων για το μέλλον μεταξύ 30 και 50% του προϋπολογισμού ε, αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας. Άρα μπορεί να μιλάμε για επικουρικότητα, αλλά ένα 30 με 50% των ε, προϋπαρχόντων προγραμμάτων υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα φαρμακευτικά σκευάσματα, για τον καπνό, για τις διασυνοριακές απειλές στην υγεία, για τους αιματολογικούς ιστούς και ούτω καθεξής. Και βεβαίως υπάρχει και η οδηγία για την για τα διασυνοριακά συστήματα υγείας. Αλλά το 30 με 50% όπως σας είπα αφιερώνεται, του, της χρηματοδότησης αφιερώνεται στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής ε, νομοθεσίας για να μπορέσουμε να έχουμε μια συνεκτική προοπτική. Ε, ο κύριος Πίτερλε μίλησε για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αν κατανόησα καλά. Αυτή είναι μια διαδικασία που δημιουργήθηκε για την ε, υποστήριξη και προώθηση των ε, αναπτυξιακών στόχων, ιδιαίτερα του στόχου 3, έτσι ώστε να μειωθούν οι χρόνιες και μεταδοτικές ασθένειες. Και το πρόγραμμα υγείας αυτό επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ε, λάβουν υπόψη αξιολογήσεις καλών πρακτικών και να τις επιταχύνουν. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που ανέλαβαν τα κράτη-μέλη. αφορούν προγράμματα κολονοσκόπησης που δεν υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη υποχρεωτικά. Πρόκειται για μία εθελούσια βάση συνεργασίας και δεύτερο, ε, η φυσική δραστηριότητα και άσκηση, φυσική άσκηση, την οποία επιβάλλει ο παθολόγος, δηλαδή την ε, ε, προβαίνει σε συνταγογράφηση αυτής της άσκησης. Αυτές είναι οι δύο πρακτικές που ακολουθήθηκαν από κράτη-μέλη με βάση το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Υγείας. Ε, μια, ένα τρίτο μέλημα αφορά την διοργάνωση εμβολιασμών. Ο κύριος Ζωρίνιο αναφέρθηκε σε αυτό. Η Επιτροπή όπως ε, ανέφερε και ο πρόεδρος Γιούνκερ στην ε, κατάσταση της Ένωσης θα προωθήσει την συστηματική, το συστηματικό εμβολιασμό του ευρωπαϊκού πληθυσμού, διότι υπάρχει ε, μια επιφυλακτικότητα από πολίτες. Αλλά έχουμε και μεγάλες δυσκολίες ως προς την, ε, τον συνεχή εφοδιασμό και ελλείψεις στα εμβόλια και επίσης ε, δεν υπάρχει ένα σωστό ε, δίκτυο φαρμακοεπαγρύπνησης στα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή θα προωθήσει μια κοινή δράση με επικεφαλή στη Γαλλία και τη συμμετοχή 20 κρατών μελών το Σεπτέμβριο για να ενισχύσουμε τη συνεργασία των κρατών μελών στον τομέα της ε, πολιτικής εμβολιασμού. Επίσης, σε σχέση με τον εμβολιασμό υπάρχει μία ε, διαδικασία δημόσιαν, δημόσιων προμηθειών που χρησιμοποιήθηκε ήδη έτσι ώστε να χορηγηθεί σε 19 κράτη-μέλη η διαδικασία και η προμήθεια πανδημικού εμβολιασμού. Άρα η Επιτροπή με 19 κράτη-μέλη προβάλλει μία κοινή ε, διαδικασία πανδημικού εμβολιασμού. Βλέπετε λοιπόν ότι η Επιτροπή προτείνει μία μελλοντική πρωτοβουλία, αλλά χρησιμοποιούμε και το ήδη προϋπάρχον πρόγραμμα υγείας για κοινή δράση στα κράτη-μέλη υπό την αιγίδα της Γαλλίας. Και είναι η πρώτη φορά που έχουμε αγοράσει μία τόσο μεγάλη ποσότητα εμπολίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, ως προς τη μελλοντική χρηματοδότηση, το πολιετές δεν έχει ακόμα εγκριθεί σε επίπεδο κομισιών. Υπάρχουν νέες ιδέες σε αυτό το αρχιτεκτόνημα, αλλά έχουμε προωθήσει αυτές τις συζητήσεις στο εσωτερικό της Κομισιόν και ένα από τα σημεία που θα ήθελα να ε, αναφέρω είναι ότι η Επιτροπή προσπαθεί να εξορθολογήσει τα προγράμματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Προσπαθούμε να μειώσουμε τον αριθμό και να, έχουμε, ε, να προβούμε σε ομαδοποιήσεις. Αυτό θα έχει πολλά πλέον εκτήματα, έτσι ώστε να μετακινηθεί το χρήμα πολύ πιο εύκολα ανάμεσα στις συνιστώσεις αυτών των ε, προγραμμάτων όπως ισχύει με την κρίση του μεταναστευτικού. Είχαμε μεγάλη δυσκολία να μεταφέρουμε κονδύλια από μία πλευρά του προγράμματος στην άλλη. Δηλαδή, όταν τα χρήματα έχουν δεσμευθεί σε μικρά προγράμματα, είναι δύσκολο να ε, γίνει ε, μεταφορά κονδυλίων. Άρα, η Επιτροπή προσπαθεί να δημιουργήσει συνέργειες και αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνονται αυτά τα προγράμματα, αλλά ομαδοποιούνται. Όπως ισχύει και με τον προϋπολογισμό. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι τομείς που εντάσσονται σε ένα κεφάλαιο. Άρα στο επόμενο πολιετές αυτό ακριβώς θα προτείνουμε είναι κάτι που διαπραγματευόμαστε, δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί δεν έχουν ακόμα ληφθεί αποφάσεις. Η κυρία Γκροστέτ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις επεξηγήσεις. Δεν είμαι πεπισμένη δυστυχώς. Κατανοώ ότι θέλουμε να απλουστεύσουμε τα πράγματα από πλευράς γραφειοκρατίας, αλλά εγώ σας μιλώ για μία πολιτική με πι κεφαλαίο. Να δείξουμε στους πολίτες ότι η πολιτική υγείας σημαίνει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη αποφασίζουν για, αποφασίζουν για το σύστημα κοινωνικής προστασίας, αλλά αν δεν παρακινήσει η Ευρώπη τα κράτη-μέλη δεν θα μπορέσει να γίνει τίποτα και θύματα θα είναι οι πολίτες. Δεν μπορώ να δεχτώ να μιλάμε για ασφάλεια τροφίμων και να μην μιλάμε για υγεία και να μιλάμε για ανθρώπινη υγεία, για υγεία των ζώων, για τα φυτά, για την ανάπτυξή τους και να μην μιλάμε για την υγεία των ανθρώπων. Εάν διαγράφουμε γραμμές του προϋπολογισμού για την ανθρώπινη υγεία και μιλάμε για ασφάλεια τροφίμων, ε, για ασφάλεια ζώων, φυτών, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Δίνουμε μία πολύχρονη μάχη για να προωθηθεί η υγεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εμείς δώσαμε και μεγάλη μάχη για να μιλάμε για Επιτροπή Περιβάλλοντος και Υγείας. Και λέω και για τους επόμενους υποψήφιους ότι δεν πρέπει να διαγραφεί το σκέλος υγεία από την Επιτροπή μας. Είναι θέμα πολιτικής ουσίας. Μας λέτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ίσως σκέφτεστε σαν εμάς, αλλά έχουμε έναν Επίτροπο Υγείας, ο οποίος είναι ενθουσιώδης, αλλά είναι απογοητευμένος γιατί δεν έχει τα μέσα να προωθήσει θέματα υγείας. Θα ήθελα η Επιτροπή μας Περιβάλλοντος και Υγείας να κινηθεί και να πούμε ότι πια φτάνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Well, um, thank you. Μάλιστα, λέει Πέτρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η σημερινή μας συζήτηση. Με τη θετική αυτή Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι αυτή την ιδέα θα την προωθήσουμε όσο μπορούμε στο πλαίσιο της Σχετικής Επιτροπής. Αγαπητοί συνάδελφοι, και έτσι ολοκληρώθηκε και οι σημερινές μας εργασίες και ξεκινάμε λοιπόν αύριο. Θα λέμε λοιπόν στις 9.30 με τους υπόλοιπους και στις 9 με τους συντονιστές.